Uh, Επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η ώρα ερωτήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρώτη ερώτηση είναι της κυρίας Μαγκίνες, αλλά την αναπληρώνει ο κύριος Χίγκινς. Ο Επίτροπος Άντορ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εξότιμη Ευρωβουλευτέ, όταν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Προστασίας ε, ε, ε, στο σημάτων ε, ε, υιοθέτησε τις ονομασίες ποιότητας, την προστατευμένη γεωγραφική ένδειξη, προστατευόμενη ονομασία προέλευσης και παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα, αντίστοιχα συστήματα ήδη υπήρχαν στα κράτη-μέλη. Η έννοια της γεωγραφικής ένδειξης ήταν γνωστή και πολλά ονόματα είχαν ήδη καταχωριστεί, πολλές ονομασίες σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλές καταχωρημένες ονομασίες σε πολλές χώρες μέλη ήδη. Βέβαια, το αυξανόμενο ενδιαφέρον στο σύστημα παρατηρήθηκε σε πολλές χώρες μέλη. Η διαδικασία καταχώρησης μιας ονομασίας ε, είναι αρκετά χρονοβόρα, κρατάει χρόνια ολόκληρα γιατί θα πρέπει να προσδιοριστούν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να εγκριθούν σε εθνικό επίπεδο. Καταρχήν και κατόπιν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα ενία έντυπα με ορισμένα χαρακτηριστικά για τις γεωγραφικές ενδείξεις ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τα εγγυημένα παραδοσιακά προϊόντα κατόπιν δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να προβληθεί μια προθεσμία εξάμεινη για την υποβολή ενστάσεων ή αντιρρήσεων. Αν δεν υποβληθούν ενστάσει, επιτρέπεται η καταχώρηση τη ονομασία. Αν όμω υποβληθούν ενστάσει, οι αφαιρόμενοι έχουν ένα εξάμεινο για να καταλήξουν σε συμφωνία. Αν δεν ε, καταλήξουν σε συμφωνία, η μόνιμη επιτροπή καταλήγει σε μια απόφαση και η διαδικασία αυτή εξηγεί και το χρόνο που χρειάζεται για την ε, υιοθέτηση μια νομοθετική πράξη. Από τη στιγμή όμω που καταχωριστεί μια ονομασία, τη χάνει ισχυρή προστασία και διεθνού αναγνώριση και υποφελείται από διάφορα επικοινωνιακά εργαλεία όπως είναι η χρήση του λογοτύπου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνέστη τις ανάγκες επιτάξεις αυτής της διαδικασίας καταχώρησης και τέτοιες προτάσεις υπε, υπευλήθησαν στο πακέτο ποιότητας προκειμένου να μειωθεί η προθεσμία εξέτασης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να μειωθεί σε δύο μήνες η προθεσμία για τις ενστάσεις. Βέβαια τα συστήματα διαφέρουν από τις διάφορες, στις διάφορες χώρες και εξαρτάται και από τις ονομασίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει κάποια κονδύλια για την πρόθεση ποιοτικών προϊόντων προκειμένου να ευαισθητοποιήσει και τους πολίτες ως προς το σύστημα προστασίας που ισχύει. Συμπληρωματική ερώτηση, ο κύριος Higgins. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ευρωπαίο Επίτροπο γιατί πιστεύω ότι η σήμανση των ποιοτικών τροφίμων είναι κάτι πραγματικά αξιέπαινο. Ο κύριος Επίτροπος επισήμενε διάφορα θέματα. Καταρχήν υπάρχουν πολλές και διάφορες προδιαγραφές. Ε, η διαδικασία είναι πολύ χρονοβόρα από τη στιγμή της αίτησης μέχρι τη στιγμή της καταχώρησης. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα γραφειοκρατίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ιρλανδία χρειάζεται πέντε χρόνια για το Υπουργείο Γεωργίας ε, από τη στιγμή της αίτηση μέχρι να καταχωρήσει την ονομασία. Χρειαζόμαστε περισσότερη σήμαση, χρειαζόμαστε περισσότερες προδιαγραφές και ελέγχους, αλλά πιστεύω ότι το χρονοδιάγραμμα που θα μπορούσε να συντομεύσει κατά πολύ. Να ακούσουμε και την ερώτηση της κυρίας Ματέρα που ζήτησε το λόγο για συμπληρωματική ερώτηση. Η κυρία Ματέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το θέμα των ποιοτικών τετροφίμων. Στην Ιταλία ε, τις τελευταίες δύο μέρες ε, ζημιά 20 εκατομμυρίων ευρώ γιατί δεν μπόρεσαν να πουληθούν κυρίως τα φασολάκια και πολλά άλλα προκυπευτικά λόγω του βακτηρίου E. coli. Το ίδιο αυτό οφείλεται στο ότι η Ρωσία ανέστηλε τι εισαγωγέ. Ε, και κατόπιν τούτου όλο αυτό το τομέα έχει γονατίσει. Και ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι είδου μέτρα προτίθεται να λάβει για να προστατεύσει αυτόν τον τομέα και τι είδου ε, μέτρα ε, πρέπει να λάβει για να μην διαδίδονται νέα που δεν είναι τεκμηριωμένα ε, και με τον τρόπο αυτό μεταφέρονται ειδήσει ε, που ε, θέτουν, που δημιουργούν πανικό σε ολόκληρους στο σύνολο του πληθυσμού. Πάντα όλα αυτά σε σχέση με το βακτήριο E. coli. Κύριε Πρόεδρε, στην πρώτη ερώτηση θα ήθελα να απαντήσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίγνωση ανάγκης επιτάχυσης ε, της νομοθετικής διαδικασίας. Έχουν υποβληθεί σχετικές προτάσεις στα πλαίσια το πακέτο ποιότητας, όπως σας είπα και στην ε, εισαγωγική μου απάντηση. Οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνουν ε, σύντμηση των προθεσμιών για την εξέταση μιας αίτησης σε έξι μήνες και μειώνουν και την προθεσμία υποβολής ενστάσεων σε δύο μήνες. Αν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αποφασίσουν να εγκρίνουν τις ε, προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα γλιτώσουμε ένα χρόνο ή τουλάχιστον δέκα μήνες για τις περισσότερες αιτήσει ε, καταγραφής. Ως προς τη δεύτερη ερώτηση, χθες συνεδρίασε το Συμβούλιο Υπουργών Υγείας, ασχολήθηκε με το θέμα αυτό, θα δοθεί κάποια συνέχεια και θα ληφθούν υπόψη ε, και τα συμπεράσματα του σημερινού Συμβουλίου Γεωργίας. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι έτοιμος να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά σίγουρα θα παρακολουθήσουμε το θέμα. Κυρία Χάρκιν, για την ίδια ερώτηση ζητήσε το λόγο για συμπληρωματική. Ναι, θα είμαι λακωνική. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν μπήκα εγκαίρως για να ακούσω την απάντηση από την αρχή. Υπάρχει ένα χαμηλό επίπεδο συνειδητοποίηση των παραγωγών σε πολλές χώρες. Ιδιαίτερα σε ορισμένε χώρες είναι τελείως, έχουν πλήρη άγνοια η Γεωργία. Θα πρέπει να αυξήσουμε λοιπόν την προσπάθεια ευαισθητοποίηση όχι μόνο του Εβραίου κοινού αλλά και των ίδιων των παραγωγών. Ο επίτροπο Άντορ. Σίγουρα είναι διαφορετική η συνειδητοποίηση του φαινομένου σε ό,τι αφορά την ανάγκη καταγραφής κάποιων ονομασιών ή της αξιοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων πάνω από 19 εκατομμύρια ευρώ δίνονται σε 15, 12 σε 15 προγράμματα προώθησης μεταξύ του 2006 και του 2010. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επανεξετάσει την πολιτική προώθηση γεωργικών προϊόντων και θα εκδώσει και σχετική πράσινη βίβλο, κάτι που θα δώσει την ευκαιρία νέας ε, εξέτασης των στόχων της πολιτικής και ανάλυσης των προσδοκιών σε ό,τι αφορά την προαγωγή ποιοτικών τροφίμων και καλύτερης διάδοσης των πληροφοριών. Σας ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση, παριθμόν 7, από τον κύριο σε σχετικά με την ανεργία των νέων. Κύριε Επίτροπε, παρακαλώ έχετε το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, η υψηλή ενεργεία ανάμεσα στους νέους είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Η έλλειψη θέσεων εργασίας ε, προφανώς ε, μπορεί να προκαλέσει την εγκατάλειψη της Ευρώπης και οι νέοι ε, θα αναγκαστούν, ε, αναγκάζονται πολλές φορές και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση να μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι λύση για περιοχές όπου υπάρχει υψηλή ανεργία νέων. Ε, σε άλλα κρατη κράτη-μέλη υπάρχει έλλειψη εργαζομένων. Αυτά προκύπτουν από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το να ενισχύσουμε την μετακίνηση των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό είναι ένα από τα μέτρα που εντάσσεται στην πρωτοβουλία ε, Ναυαρχίδα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να σας αναφέρω και ορισμένα παραδείγματα. Ε, η, μετακίνηση, η ελεύθερη μετακίνηση των νέων προάγεται με ένα νέο πρόγραμμα το οποίο εισήχθη με τη δική σας υποστήριξη και του Συμβουλίου. Στόχος έχει το πρόγραμμα αυτό να βοηθήσει τους νέους να βρουν θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και να βοηθήσουν βοηθήσει τους εργοδότες ε, να προσλαμβάνουν νέους ε, μετακινούμενους εργαζόμενους ε, προσφέρονται συμβουλές για την αναζήτηση εργασίας αλλά και οικονομική υποστήριξη μέχρι και χίλια ευρώ αυτό προσφέρεται σε νέους αλλά μάλλον σε εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν νέους. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι τέσσερις μήνες μετά τη γενική τους εκπαίδευση την χάνουν και ειδική κατάρτιση. Στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ολλανδία, όπως πολύ σωστά επισημαίνει και ο κύριος Ευρωβουλευτής, η ενεργεία των νέων είναι σχετικά χαμηλή. Αυτό οφείλεται εν μέρη στο ότι υπάρχει πολύ καλή επαγγελματική κατάρτιση ε, σε αυτά τα κράτη ε, που ε, διευκολύνει την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας το ανακοινωθέν του 2010 σχετικά με την ε, καλύτερη συνεργασία για την επαγγελματική κατάρτιση για την περίοδο 2011-2012 αυτό είναι ένα σημαντικό ευρωπαϊκό επίτευγμα. Ε, προβάλλει τους στόχους και εντοπίζει ε, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στην επαγγελματική κατάρτιση και επιπλέον καθιστά τους νέους περισσότερο ενδιαφέροντες για την αγορά εργασίας. Να προσθέσω και κάτι άλλο στην απάντησή θα ήθελα να επισημάσω τη χρησιμότητα της ε, εκστρατείας ε, εργασίας που ξεκίνησε στη Βουδαπέστη τον Απρίλη και αυτό, αυτή η εκστρατεία απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε νέους. Εμείς προσφέρουμε πληροφορίες για να εμπνεύσουμε τους νέους να ανοίξουν τη δική τους ε, τη δουλειά. Μέχρι τώρα υπάρχει κάποια επιτυχία και θα συνεχιστεί ελπίζουμε η επιτυχία αυτή μέχρι το τέλος του 2012 που θα ολοκληρωθεί και η εκστρατεία εκστρατεία. Ελπίζω αυτά που σας είπα ε, να συνοδευτούν και από αποτελεσματικά μέτρα στα κράτη-μέλη. Πρόεδρος, ε, κύριε Higgins ε, και μετά Ζέμκλερ και Τίκαου. Δυστυχώς δεν μπορώ να δώσω το λόγο στον κύριο Παπα-Νικολάου και στην κυρία Γκουτιέρε, γιατί επιτρέπονται μόνο τρει συμπληρωματικέ εργασίε. Ο κύριο Χίγκιν. Κύριε Πρόεδρε, τα ε, στοιχεία τρομάζουν. Οι χώρε τη Βαλτική, η Ιρλανδία, η Ελλάδα και η Σλοβακία, 30%, η Ισπανία 40% και στη δική σα τη χώρα ένα εκατομμύριο άνθρωποι κάτω τη ηλικία των 25 ετών με καμία προοπτική εργασία. Ε, στην Ιρλανδία ε, πολλοί νέοι θα μεταναστεύσουν. Ε, θα ήθελα η μετακίνηση η ελεύθερη να είναι η απάντηση, όμως ε, δεν ισχύει αυτό. Εκείνο που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι να εστιάσουμε την προσοχή μας στο γεγονός ότι στην Ευρώπη έχουμε γυράσκοντα πληθυσμό. Δεν μας επιτρέπεται αυτή η πολυτέλεια της ε, διαρροής εγκεφάλων. Χρειαζόμαστε τους νέους, πρέπει να τους κρατήσουμε εδώ, μέσα σε προγράμματα σαν αυτά που αναφέρεται στις τρεις χώρες, Γερμανία, Ολλανδία και Αυστρία. Χαιρετίζω λοιπόν το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτείνει πρωτοβουλίε στα κράτη-μέλη. Βέβαια, ορισμένα κράτη-μέλη χρειάζονται οικονομική βοήθεια για την κατάρτιση για να κρατήσουν του νέου. Γιατί πιστεύω ότι αντί να ε, τροφοδοτείται η αγορά εργασία Ευρωπαϊκή Ένωση, τροφοδοτείται η αγορά τη Αυστραλία και άλλων κρατών. Πρόεδρος, να σας υπενθυμίσω ότι 30 δευτερόλεπτα έχετε για τις συμπληρωματικέ ε, επόμενη παρατήρηση. Ε, Ο κύριος Ζέμκε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και έχω μια ερώτηση προς τον Επίτροπε, αλλά κάπως διαφορετικού είδους. Μιλήσατε κύριε Επίτροπε για τις διάφορες ε, δραστηριότητες και πρωτοβουλίες για τη μείωση της ανεργίας, αλλά δεν είπατε ούτε κουβέντα για το γεγονός ότι ένας αποτελεσματικός τρόπος θα ήταν οι χώρες μέλη να λάβουν υπόψη και τα προσόντα και τις δεξιότητες που, ε, ανακτά, που αποκτά κάποιος σε άλλες χώρες. Τι θα γίνει με αυτό, με την αναγνώριση δηλαδή των δεξιοτήτων που αποκτούνται σε άλλες χώρες. Η κυρία Τσικάου. Ευχαριστώ. Η υψηλή ενεργεία των νέων δείχνει ότι οι επενδύσεις ορισμένων χωρών στην παιδεία ε, έχουν πάει χαμένες γιατί οι νέοι δεν βρίσκουν δουλειά και ξαναγκάζονται να αποδημήσουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεδομένου το επίπεδο της εγκατάλειψης της σχολικής φίτησης έφτασε από 16% μέχρι 40% σε ορισμένες χώρες όπως η Πορτογαλία. Ποιο θα είναι το επίπεδο ενεργείας των νέων μέσα σε μία 20 ετία και πώς θα αναχαιτήσουμε αυτές τις ανησυχητικές τάσει. Ε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, στην απάντησή μου επισήμανα τα μέτρα τα οποία ε, ήδη αναφέρονται στην ε, στρατηγική Ευρώπη 2020. Και είπα ότι τα μέτρα αυτά ήδη εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη-μέλη ε, μέσα από αποτελεσματικά προγράμματα που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι αλήθεια ότι αυτό είναι ένα οριζόντιο θέμα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχουν και άλλες ε, πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, πολύ σημαντικές ε, προτάσεις, παραδείγματο χάρη συμπεριλαμβανομένων και των συστάσεων που απευθύνονται σε ειδικά σε συγκεκριμένες χώρες. Αυτή δημοσιεύτηκε σήμερα και αναφέρονται ότι είναι απαραίτητο να μεταρρυθμιστούν οι εκπαιδευτικές πολιτικές και να βελτιωθεί η απόδοση των συστημάτων κατάρτισης σε ορισμένα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη διασύνδεση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά οι δυνατότητες απασχόλησης των νέων σε αρκετά κρατημέλη, μεταξύ αυτών και στην Ισπανία, όπου η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και όπου η μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος είτε καθυστέρησεται, ε, αγνοήθηκε τα τελευταία χρόνια. Ε, αναφερθήκαμε και στην ε, πράξη της ενιαίας αγοράς μεταξύ άλλων έχει ως στόχο να προάγει την αναγνώριση πτυχίων και δεξιοτήτων. Με τον τρόπο αυτό η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας θα καταστεί περισσότερο διαφανής, αποτελεσματική, θα υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες από ό,τι κατά το παρελθόν. Είναι εξάλλου σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι πάρα πολλές ενέργειες στηρίζονται από το δημοσιονομικό ε, μέσο, τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι κυρίως εδώ ε, στο Κοινωνικό Ταμείο και στην ε, νέα μικροχρηματοδοτική δυνατότητα που ενισχύει ε, προγράμματα ε, επιχειρηματικότητας. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό εργαλείο. Και θέλω να πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα στηρίξει τις προτάσεις της Επιτροπής στο πρόγραμμα αυτό. Και ερχόμαστε, ευχαριστώ, στην επόμενη ερώτηση του κυρίου Παπα-Νικολάου, μετανάστευση και Σέγγεν, υπαριθμών 8. Θα απαντήσει η κυρία Μάνστομ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Η ερώτηση του κυρίου Παπα-Νικολάου, όπως και επόμενες ερωτήσεις, ασχολούνται με τα διάφορα θέματα ε, του Σέγγεν και την κρίση, τη μετανάστευση και τις πιέσεις που υφίσταται το Σέγγεν. Θα απαντήσω σε εσά πρώτα κύριε Παπα-Νικολάου. Το έχουμε συζητήσει προηγουμένως, ε, πριν συζητούσαμε την έκθεση του κυρίου Κοέλιο και την ανάγκη να διαφυλάξουμε το Σέγγεν που είναι από τα πιο όμορφα επιτεύγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι πολύ σημαντικό δικαίωμα και πολύ ε, σημαντική ενσάρκωση της ευρωπαϊκής ιδέας και ε, κάθε χρόνο ένα δισεκατομμύριο, 250 εκατομμύρια ε, πολίτες ταξιδεύουν ως τουρίστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τονώνεται έτσι και η εσωτερική αγορά. Είναι τεράστια προτεραιότητα και για την Επιτροπή και για μένα προσωπικά αυτό. Πρέπει να σας πω και πάλι ότι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ενίσχυση του ΣΕΝΓΕ, να βελτιωθεί ε, ε, επαλήθευση όπως δεσμευτήκαμε πριν τα Χριστούγεννα να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να δούμε ποια είναι τα εργαλεία και ενδεχομένως να υιοθετήσουμε και ένα μηχανισμό για μια κοινή κοινοτική ανταπόκριση σε έκτακτες περιστάσεις. Ε, ας πούμε ε, όταν έχουν θέματα τα κράτη-μέλη για τα εσωτερικά σύνορα. Θα πρέπει να είναι προληπτική η ε, προσέγγιση. Κοινός μηχανισμός για να διατηρηθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά ε, με συνοδευτικά μέτρα για να διαφυλαχθεί ένας χώρος χωρίς σύνορα. Αυτό ε, θα γίνει με επιτόπου ε, επισκέψεις στα κράτη-μέλη με ελέγχους που μπορεί να καταλήγουν και σε συστάσεις για άμεση δράση με προθεσμίες στα κράτη-μέλη για να τις εφαρμόζουν. Η αύξηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών θα μειώσει ε, και τη λήψη μονομερών μέτρων, την προσφυγή σε τέτοιες καταστάσεις μονομερός από κράτη-μέλη για επαναφορά των ελέγχων στα σύνορα ή αστυνομικά μέτρα. Το Σέγγεν είναι ένα ένα πνεύμα αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης. Είναι σημαντικό να είναι συγκεκριμένη η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις χώρες που πλήττονται ιδιαίτερα από τις μεταναστευτικές πιέσεις και από πρόσωπα που χάνουν και χρειάζονται διεθνή προστασία. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Ε, βοήθεια, Frontex ε, στα εξωτερικά σύνορα όταν δέχονται μεγάλες πιέσεις. Έχουμε δει πρόσφατα ε, την επέμβαση Rabbit στα ελληνοτουρκικά ε, ε, ταχεία επέμβαση ε, και την επιχείρηση Ερμής. Επίσης θα πρέπει καθημερινά να συνεργάζονται τα κράτη-μέλη για τη φύλαξη των συνόρων και αυτό είναι και το ευρωπαϊκό αντίστοιχο σύστημα το οποίο σιγά σιγά εξελίσσεται από το 2008 και θα κάνει νομοθετική πρόταση φέτος ακόμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης μπορούμε να επιδείξουμε την αλληλεγγύη και με με ε, οικονομικό τρόπο. Υπάρχει ένα πλαίσιο, ένα πρόγραμμα φέτος που λαμβάνει υπόψη του τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και έχουμε και ε, χρηματοδοτικό μηχανισμό για να βελτιώσουμε τη διαχείριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ενισχύσουμε και πάλι την αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών. Βεβαίως τώρα έχουμε ε, μια μεγάλη διαδικασία διαβούλευσης, έχουμε και δημοσιονομικούς περιορισμούς, αλλά μπορείτε να υπολογίζετε σε μένα ότι θα υπάρξουν χρήματα σε αυτό το ταμείο και για το μέλλον. Τα κράτη-μέλη εκείνα που εκτίθεται περισσότερο στις μεταναστευτικές πιέσεις και ε, βρίσκονται και στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης θα πρέπει να δέχονται οικονομικές αποζημιώσεις για τα καθήκοντα που ασκούν προς όφελος όλου του χώρου Σέγγεν με δίκαιη κατανομή του άχθους ε, υποστηρίζουν τα κράτη-μέλη ε, ακριβώς ε, που δέχονται μεγάλες πιέσεις και μεγάλο αριθμό ατόμων που χρειάζονται νομική προστασία διεθνή. Βεβαίω, οποιαδήποτε απόφαση θα εξαρθεί από τα κράτη-μέλη και από το Συμβούλιο. Τα κράτη-μέλη ακόμα δεν έχουν υποστηρίξει μια τέτοια προσέγγιση έτσι γενική με μια αξιόλογη ε, εξαίρεση το πιλωτικό πρόγραμμα ε, επανεγκατάστασης ε, σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκείνων που ζήτησαν προστασία στη Μάλτα. Πριν από ένα μήνα μάλιστα διοργάνωσα και μία διάσκεψη δωρητών και χαίρομαι που πάνω από 300 ήταν οι προσφορές από χώρες και από συνδεδεμένες χώρες ε, και στο μέλλον θα προσθεθούν και άλλοι. Αυτό είναι η αλληλεγγύη στην πράξη συγκεκριμένα και θέλω να ευχαριστήσω τις χώρες αυτές και ελπίζω στο μέλλον να βοηθήσουν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη που μακρηγόρησα αλλά αφορά και επόμενες ερωτήσεις όπου θα είμαι πιο σύντομη. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Κύριε Παπα-Νικολάου πρώτα και μετά ο κύριος Λιβία. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και συμφωνώ απολύτως μαζί σας, όπως νομίζω συμφωνεί και το Κοινοβούλιο μας. Αυτό φάνηκε και προηγουμένως στη συζήτηση για την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Την ίδια στιγμή όμως, ξέρετε καλά ότι στο Συμβούλιο υπάρχει ζήτημα ομοφωνίας για το θέμα της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Μιλήσατε για εμπιστοσύνη. Ναι, θέλουμε να οικοδομούμε συνεχώ την εμπιστοσύνη. Η Δανία αποδέχεται όμω τη δήλωσή σα, αυτή με την επιλογή που έχει κάνει. Τοποθετηθήκατε επίση για, τον το νέο μηχανισμό. Εν ώψη και τη Συνόδου Κορυφής, η συζήτηση αυτή για το μηχανισμό ενισχύει την αντίληψη για την εμπιστοσύνη που ούτω ή άλλω θυμίζω ότι στο, στον κώδικα Σέγγεν στο άρθρο 23 υπάρχει μηχανισμό για εξαιρετικέ περιστάσει ή τελικά προκαλεί νέα ανησυχία στα κράτη μέλη και σε όσα κράτη βρίσκονται στον χώρο Σέγγεν. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. 30 δεύτερα είναι η συμπροματική. Ο κύριος Λαβία παρακαλώ. 32 32η. Señor Κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τον επόμενο μήνα θα διατυπώσει την πρόταση του νέου πολιτέ σε δημοσιονομικού πλαισίου ε, για το 2013 στο 2020. Έτσι λοιπόν, ε, πέρα από τη Frontex που αναφέρατε, τι άλλου είδου δράσει προτίθεται η Κομισιόν να χρηματοδοτήσει για να στηρίξει τα κράτη-μέλη τα οποία πλήττονται από θέματα ασύλου και για να μπορέσει στο μέλλον να αποτρέψει οικονομικού μετανάστε. Με άλλα λόγια, είδου είδους ενέργειες προτίθεστε να χρηματοδοτήσετε μέσα από την πολιτική γειτονία ε, για να μπορέσετε να παρεμποδίσετε μεταναστευτικές ροές που προβλέπονται για τους επόμενους μήνες και για τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπος, σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, η εμπιστοσύνη δεν ε, επιβάλλεται, δεν διατάσσεται, εμπνέεται και κερδίζεται. Και μπορούμε να βελτιώσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μελών με ε, καλύτερη διαχείριση και εποπτεία του Σέγγεν και ε, να Έχουμε έναν εξάρτητο μηχανισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο κοινοτικό, όχι το σημερινό σύστημα που είναι αξιολόγηση μεταξύ ίσων ή ομοτήμων, αυτό το peer review. Να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύνολο εργαλείων για να μπορούμε να βοηθούμε τα κράτη-μέλη που ε, αντιμετωπίζουν ε, δυσκολίες και ελπίζω να αυξηθεί η εμπιστοσύνη. Απαντώ στον κύριο Λαβία και προς τον κύριο Παπα-Νικολάου. Ε, δεν έχω αριθμητικά στοιχεία να σας δώσω, αλλά θέλουμε να αυξήσουμε και την ανεξαρτησία και τους πόρους και τη στελέχωση και τον εξοπλισμό του Frontex, ε, να έχουν τα κράτη-μέλη πρόσβαση σε διάφορα ταμεία για τη μετανάστευση με απλοποίηση και για τα ε, σύνορα και για την ένταξη και για το άσυλο κτλ. Βεβαίως θα πρέπει να γίνεται πάντα η διάκριση μεταξύ λάθρων μεταναστών και μεταναστών ε, που χρειάζονται διεθνή προστασία. Όπως γνωρίζετε τώρα το Συμβούλιο διαπραγματεύεται με το Κοινοβούλιο για αυτό το πρόγραμμα επανεγκατάστασης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να κοιτάξει τι δυνατότητες υπάρχουν για χρηματοδότηση πολλών τέτοιων προγραμμάτων και σε σχέση με την άμεση γειτονία ε, στη Μεσόγειο ε, με την εταιρική ε, σχέση μπορούμε να κοιτάμε όλες τις πτυχές και την νόμιμη μετανάστευση και την παράνομη και το άσυλο και την προστασία. Όλα αυτά χρειάζονται πολιτική βούληση, ορισμένα επιπλέον μέσα και σας διαβεβαιώ ότι είναι στη δική μου αρμοδιότητα θα φροντίσω να προωθηθεί. Ευχαριστώ. Ωραία, περνάμε στην ένατη ερώτηση του κύριου Πόσελτ για το καθεστώς θεωρήσεων για το κοσυφοπαίδιο. Η Επίτροπος. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, κύριε Πόσελτ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή παρακολουθεί εκ του συνεγγύς όλα τα βήματα που πραγματοποιούν οι αρχές του κοσυφοπεδίου προκειμένου να στρέξουν οι προϋποθέσεις για την απελευθέρωση για το διαλόγο για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Δύο είναι τα εκκρεμή βασικά θέματα για να ξεκινήσουμε το διάλογο αυτό. Ε, σωστή επανεισδοχή και πολιτική επανένταξη που θα τηρεί τι ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ. Η εφαρμογή του, του νόμου για την επανεισδοχή και διμερεί ε, συμφωνίε επανεισδοχή μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και των μελών θα πρέπει να συνεχιστούν. Ε, πραγματοποιήθηκαν δύο αποστολέ αξιολόγηση, πέρυσι τον Ιούνιο και πέρυσι τον Δεκέμβριο στο Κωσυφοπέδιο, για να εκτιμηθεί η εξέλιξη των πραγμάτων σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ε, απελευθέρωση των θεωρήσεων. Πρόοδος έχει συντελεστεί, αλλά θα πρέπει να συνεχιστεί. Συνεχίζουμε το διάλογο με την κυβέρνηση του Κωσυφοπεδίου, προκειμένου να την βοηθήσουμε για να ε, ολοκληρώσει τις τελευταίες εκκρεμότητες και να σημειωθεί πρόοδος και σε περιφερειακό επίπεδο. Γίνονται τακτικές ε, επικαιροποίησεις από τις αρμόδιες αρχές. Έχουμε συναντήσει με τους αρμόδιους υπουργούς και από τη στιγμή που θα είναι έτοιμη η κατάσταση και έτοιμο το κοσυφοπαίδιο θα πραγματοποιήσουμε νέα αποστολή για να δούμε τι περαιτέρω βήματα θα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσει ο διάλογος απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Δεν έχουμε ε, φτάσει ακόμη στο πέρας της διαδικασίας, αλλά σημειώθηκε πρόοδος και έχουμε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση προκειμένου να τη βοηθήσουμε για να πραγματοποιήσει περαιτέρω πρόοδο. Κύριος Πόσελτ. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ καλή σας απάντηση. Θέλω μόνο να ρωτήσω το εξή. Θεωρείτε ότι είναι πιθανό η αποστολή αυτή ε, φέτο ε, να μεταβεί ε, στο 25, μήπως δεν μπορείτε να το προβλέψετε τώρα και θεωρείτε ότι είναι τόσο σημαντικό μια τόσο μικρή χώρα που τη στηρίζουμε με τόσα πολλά χρήματα να μην μπορεί να στείλει τους ανθρώπους στην Ευρώπη. Είναι αντιφατικότερο να τους κλείνουμε εκεί. Ξέρω ότι θέλετε να ανοίξουν τα σύνορα, αλλά θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστικό αυτή η αποστολή να λάβει χώρα ήδη κατά την Πολωνική Προεδρία. Συμφωνώ απόλυτα και στερνίζομαι τις φιλοδοξίες σας ε, να αποφύγουμε να γίνει ένας απομονωμένος θύλακας στο κοσυφοπαίδιο μέσα σε μια ευρύτερη περιοχή. Προσπαθούμε σταδιακά να άρουμε τους φραγμούς ε, των θεωρήσεων. Δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε το κοσυφοπαίδιο, αλλά εναπόκειται και στη δική τους προσπάθεια. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε και όταν μας πει ότι είναι έτοιμο το κοσυφοπαίδιο και πραγματοποιήσει τις υποχρεώσεις του θα στείλουμε την επόμενη επιστολή. Δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια. Η αποστολή θα πραγματοποιηθεί μόλις μας καλέσει το κοσυφοπαίδιο και πει ότι είναι έτοιμο. Ευχαριστώ. Δέκατη ερώτηση του κυρίου Μίτσελ για την καταμέτρηση της χρήσης του διαδικτύου από εγκληματίες. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Thank you very much, Mr. President. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, αγαπητά μέλη, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο είναι μια αυξανόμενη απειλή γιατί μετακινείται όλο και πιο εύκολα και οι αναλύσεις δείχνουν ότι το οργανωμένο έγκλημα εμπλέκεται στο έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν τα παρακολουθεί όλα αυτά εκ του σύνεγγες ε, για να ε, προλάβει επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Έχουμε χάρτες πορείας, ε, στόχους, αναφέρονται αυτοί σε σχετικά έγγραφα, έχουμε την ατζέντα και έχουμε και την δική μας την στρατηγική στην οποία το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αντιμετωπίζεται ως μία από τις προτεραιότητές μας για το μέλλον. Πέρυσι ε, καταθέσαμε και δύο νομοθετικές προτάσεις, η μία το Μάρτιο, μία οδηγία ε, για την εκμετάλλευση των παιδιών επιγραμμικά. Ξέρω ότι συζητείται τώρα αυτή η οδηγία και κατόπιν μία πρόταση για αντιμετώπιση επιθέσεων ε, στον κυβερνοχώρο. Αυτό έγινε το Σεπτέμβρη. Ε, το συζητήσατε και εσείς και το συζητάτε με το Συμβούλιο και γνωρίζω ότι σημειώνεται πρόοδος. Βέβαια, στόχος είναι να υπάρξει ευρωπαϊκή νομοθεσία γιατί είδαμε ότι υπάρχουν απειλές και συμπεριλάβαμε και πρόστιμα, κυρώσεις ε, για κακόβουλες ε, πράξεις. Η διεθνή συνεργασία είναι επίση το κλειδί για να αντιμετωπιστεί το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και γι' αυτό συνεργαζόμαστε με άλλου εταίρου σε διεθνέ επίπεδο. Υπάρχει ομάδα εργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ΗΠΑ που συστήθηκε το Νοέμβριο του περασμένου έτου, όπου στην ομάδα αυτή, ε, η ομάδα αυτή ε, συναντήθηκε πολλέ φορέ ε, και θα καταθέσουν την πρόοδό του στην επόμενη συνάντηση κορυφή του Νοεμβρίου. Εξάλλου θέλουμε να υπάρχει ένα κυβερνοκέντρο όπου θα συντονίζονται οι προσπάθειε καταβάλλονται στα διάφορα κράτη-μέλη. Το κυβερνοέγκλημα επηρεάζεται άμεσα, άμεσα από την ταχεία τεχνολογική πρόοδο. Προκύπτουν νέα επιχειρησιακά μοντέλα, αλλά και η δυνατότητα, η ε, δίωξη του εγκλήματος να αντιμετωπίσει το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Γιατί πλέον ε, το έγκλημα αυτό επεκτείνεται όλο και περισσότερο και ω εκ τούτου ε, χρειαζόμαστε να έχουμε τα απαραίτητα συστήματα να ανταλλάσσουμε πληροφορίες για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Αν θεωρούμε ότι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος χρησιμοποιούν όλο και το περισσότερο το διαδίκτυο, το ίδιο ισχύει και για τη διεξή τους το επιγραμμικό έγκλημα ε, θα πρέπει να ε, συντονίζεται με διάφορους μηχανισμούς. Πριν από 10 χρόνια η σύμβαση της Βουδαπέστης του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο υπογράφηκε τότε η σύνταξη αυτή. Έχουν περάσει 10 χρόνια αλλά δεν έχει επικυρωθεί η σύμβαση αυτή από όλα τα κράτη-μέλη και γι' αυτό εμείς πιέζουμε να ε, έχει επικυρωθεί όταν θα έχουμε την δεκαετή επέτειο από ε, τη συμφωνία αυτής της χώρας έτσι ώστε όλα τα κράτη να δεσμευτούν να αντιμετωπίσουν το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και την κυρία Επίτροπο για την απάντησή της. Ε, ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι ε, που μέσα από το διαδίκτυο ε, έχουν εγκληματικές επιχειρήσεις, πορνεία, εμπόριο όπλων, λαθρέα εισαγωγή ανθρώπων μέσα από τα σύνορα, δολοφονίες, ληστείες, ένοπλες ληστείες και πάρα πολλά άλλα όλα αυτά ε, γίνονται μέσα από την κατάχρηση του συστήματος. Η Europol και η ε, παροχή, ε, αν συντονιστούν, σίγουρα μπορούν να εντοπίσουν ορισμένους από αυτούς τους δράστες, γιατί αυξάνονται όλο και περισσότερο. Καλό λοιπόν την Κομισιόν να εξετάσει κάποια συγκεκριμένα μέτρα για συντονισμένη απάντηση σε αυτά που πράττουν οι άνθρωποι αυτοί μέσα από το διαδίκτυο. Ε, Ευχαριστώ. Ε, το εύρος, η βαρύτητα των ε, επιθέσεων στο κυβερνοχώρο είναι όλο και μεγαλύτερη, με θύματα διάφορους οργανισμούς και πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει τη δράση της και τη στρατηγική της για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. στα πλαίσια της διεύρυνσης της εντολής ε, του εν λόγω μηχανισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι προτίθεται να κάνει, η Επίτροπος. Σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, το ε, καθημερινό έγκλημα και αυτό γίνεται μέσα από το διαδίκτυο, γιατί αυτό χρησιμοποιείται το διαδίκτυο. Αλλά υπάρχουν και νέε μορφέ εγκλήματο που διευκολύνονται από το διαδίκτυο, όπω ε, οι δόλοι χειρισμοί, η φαρπαγή στοιχείων και ε, στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Έχουν λοιπόν υπάρξει πολλέ επιθέσει δικέ μα εναντίον αυτών των συμμοριών. Του έχουμε εντοπίσει, Ας πούμε, αυτού που ασχολούνται με την παιδική πορνογραφία αλλά και με την παράνομη διακίνηση ανθρώπων και το λατρεμπόριο. Οι ομάδε τη ε, Europol είναι εξειδικευμένε και ασχολούνται με αυτό. Βέβαια πρέπει να συνδυάσουμε όλα τα κέντρα ε, που υπάρχουν και εκδίδουν συναγερμού. Ε, πρέπει να ανταλλάσσουμε πληροφορίε, να συνεργαστούμε περισσότερο με τι ιδιωτικέ εταιρείε για να βρούμε τι λύσει σε κάποιο βαθμό. Επίσης ε, σχεδιάζουμε να ε, καταρτήσουμε μελέτες ε, σκοπιμότητας, να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κέντρο αντιμετώπισης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Σύντομα να υπάρχει αυτό. Θα είναι ένα κέντρο που θα εκδίδει συναγερμό και θα συντονίζει τα διάφορα κέντρα για την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος που ήδη υπάρχουν. Ε, θέλουμε να συνεργαστούμε με τις εθνικές αρχές ε, και αυτές ε, καλούνται να κάνουν ό,τι μπορούν για να αντιμετωπίσουν το όλο και αυξανόμενο αυτό έγκλημα. Ευχαριστώ πολύ και ερχόμαστε ερωτήσεις 11 και 12 της Βαρόνης Λάτσπορτ και της κυρίας Μαρίας Ελένης Κοπά με θέμα το Σέγγεν και την εφαρμογή της συνθήκης. Ευχαριστώ, Επίτροπος. Θα απαντήσω από εκείνο και στις δύο ερωτήσεις γιατί σχεδόν ταυτίζονται και ε, μιλούν για τη διατήρηση και τη μεταξέλιξη του Σέγγεν σε μια ε, περίοδο μεταναστευτικής κρίσης. Ήδη απάντησα εν μέρη, απαντώντας τον κύριο Παπα-Νικολάου, αλλά και αυτά τα στοιχεία θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη, αυτά που είπα προηγουμένως. Το θέμα της κυρίας Λάτφορτ ανησυχεί για ε, τις διαδικασίες και τις διαπραγματεύσεις και ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κατά προτεραιότητα προσφυγή κατά των μελών που παραβιάζουν το Σέγγεν. Κοιτάξτε, ε, θα πρέπει να είμαι ξεκάθαρη. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε παραβίαση των κανόνων του Σέγγεν. Αλλά το ένα δεν αποκλείει το άλλο και παράλληλα θα έχουμε μια άλλη διαδικασία. Εμείς ε, είμαστε οι θεματοφύλακες του κοινοτικού νόμου και θα εξακολουθήσει να ε, φροντίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι πάντες να δέχονται και να εφαρμόζουν το Σέγγεν. Το θέμα είναι η φυστάμενη νομοθεσία. Η φυστάμενη νομοθεσία μπορεί να αντιμετωπίσει ε, στη συντριπτική πλειονότητά του τα θέματα. Μπορεί να υπάρχουν χωρί την ερμηνεία αλλά στην εφαρμογή και τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έρχεται σε επαφή, θα διαβουλεύεται με τι εν λόγω χώρε και θα διευκρινίζει του κανόνε με συστάσει ή κατευθυντήριε γραμμέ. Για να βεβαιωθούμε ότι εφαρμόζεται σωστά ο κοινοτικό νόμο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέτρα που έχει στη διάθεσή τη και μεταξύ αυτών και προσφυγή επί παραβιάση όταν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Ταυτόχρονα ε, θα έχουμε και προληπτικά μέτρα για να αποφύγουμε διαδικασίες επί παραβάση. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν ε, διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων για την εκπόνηση ε, ενός συστήματος αξιολόγησης του Σέγγεν πιο αποτελεσματικού για να δούμε ε, αν και πότε θα ολοκληρωθεί αυτός ο μηχανισμός για να δημιουργηθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη και να ε, γίνεται σωστά εφαρμογή των κανόνων. Σε ό,τι αφορά τα σχέδια της δανικής κυβέρνησης για την επαναφορά συνοριακών ελέγχων, όπως ρωτάει η κυρία Κοπά, βεβαίως θα γνωρίζετε ότι αμέσως απίφθηνε επιστολή στον Δανό Πρωθυπουργό ο κύριος Μπαρόσο, λέγοντας ότι η πρώτη ανάλυση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, οδήγησε σε μεγάλες αμφιβολίες κατά πόσο ε, ανταποκρίνεται η Δανία στις υποχρεώσεις της απέναντι στο κοινοτικό νόμο και στο διεθνές δίκαιο. Τόνισε ο κύριος Μπαρόσο ότι δεν μπορούν συστηματικά ε, να επαναφέρουν συνοριακούς ελέγχους, είτε πρόκειται για ε, ε, πρόσωπα είτε πρόκειται για εμπορεύματα. Αναλύουμε τις πληροφορίες που ζητήσαμε από τη Δανία και θα ακολουθήσει απόφαση για περαιτέρω δράση. Επίσης, η κυρία Κόπα ρωτάει αν θα προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αναθεώρηση της αρχής της αποκλειστικής αρμοδιότητας του κράτους πρώτης παράνομης εισόδου Ε, αυτό είναι ειδικό κανόνα από το Δουβλίνο, ο κανονισμό του Δουβλίνου ορίζει ότι η αρμόδια χώρα για να εξετάσει μια αίτηση ασύλου ε, ε, είναι η πρώτη χώρα, δεν είναι κάτι όμως που έχει να κάνει με την παράνομη μετανάστευση αυτό. Στη πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού του Δουβλίνου παραμένει άθικτος αυτός ο κανόνας. Θα πρέπει η χώρα της πρώτης εισόδου να ελέγχει την αίτηση ασύλου. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μάιο του 2009 υποστήριξε συντριπτικά ε, αυτή την πρόταση, καθώς επίσης και η Επιτροπή Ελευθεριών πέρυσι το Νοέμβριο. Το επιβεβαίωσε. Η Βαρόνι Λάτφορτ για την πρώτη συμπληρωματική ερώτηση, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Επίτροπο και βεβαίω χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω να τονίζετε και πάλι τη σημασία που αποδίδεται στη διατήρηση του χώρου του Σέγγεν. Ξέρω ότι είστε πολύ ειλικρινείς, αλλά ανησυχώ, γιατί ε, παρόλα αυτά δημιουργήθηκε η εντύπωση την περασμένη εβδομάδα έγραψα ένα άρθρο Financial Times που έλεγε ότι διαλύεται και το Σέγγεν όπως και η Ευρωζώνη έχουν τη λανθασμένη εντύπωση οι άνθρωποι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάρα πολύ χαλαρή απέναντι στα όσα συμβαίνουν και στην επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στα ιστορικά σύνορα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει το θεσμικό της ρόλο, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται στην πράξη, στην επίδειξη αποφασιστικότητας και ζήλου να προχωρήσετε. δεν έχω ακούσει για την επιστολή της Κοπεχάκης, α πούμε να το συζητάνε στη Ρώμη, στο Παρίσι. Κυρία Κοπά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την απάντησή σας, την καθαρή απάντηση για το θέμα του Σέγγεν, καθώς και την αναφορά που κάνατε σε προηγούμενη ερώτηση για την, το μέτρο ανακατανομής μεταναστών στα κράτη-μέλη ανάλογα με πληθυσμιακά, οικονομικά, γεωγραφικά κριτήρια σε κάθε περίπτωση στο θέμα του κανονισμού δουβλίνου ii θέλω να πω ότι σήμερα για ορισμένες χώρες όπως είναι η χώρα μου η ελλάδα που αποτελούν τα εξωτερικά σύνορα της ένωσης και όπου πραγματικά είναι χώρες που δέχονται περίπου το 90% των μεταναστών που μπαίνουν στην ελλάδα ο κανονισμός δουβλίνου 2 δεν είναι ανεκτός. δεν είναι κάτι που μπορούν να το αντέξουν οι πληθυσμοί δεν είναι κάτι που μπορούν να το αντέξουν οι χώρες. επομένως από τη δική μου πλευρά από τη δική μας πλευρά είναι ένα πάγιο αίτημα για αναθεώρηση τουλάχιστον υπό το φω των νέων εξελίξεων. Σας ευχαριστώ. παπα Επίτροπε, αναφέρατε και προηγουμένως την έμφαση στην έννοια της αλληλεγγύης στη δίκαιη κατανομή των βαρών και ε, πολύ σωστά μας υπενθυμίσατε ότι επίκυνται οι διαπραγματεύσεις για την επανεγκατάσταση προσφύγων από τρίτες χώρες. Ε, είχατε ανακοινώσει και πέρυσι ότι αναμένουμε και το νέο πρόγραμμα για την εσωτερική επανεγκατάσταση. θα ήθελα να μας πείτε αν είμαστε κοντά στο να το ανακοινώσει η επιτροπή. και δεύτερον σε ό,τι αφορά το δουβλίνο 2 και συμπληρώνω σε αυτό που είπε η συνάδελφος η κυρία κοπά η γαλλία ανέστειλε τις επιστροφές στην ελλάδα η γερμανία το ίδιο. το ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας καταδίκασε για συγκεκριμένους λόγους και για το δουβλίνο 2 και τη λειτουργικότητα αυτού. τι άλλο πρέπει να συμβεί για να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει αμέσως να αλλάξει το δουβλίνο 2 όπως ζητάει το κοινοβούλιο μας. Σας ευχαριστώ. παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Λυπάμαι αν έχει δοθεί εσφαλμένη εντύπωση για το τι φρονεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Σέγγεν. Το τελευταίο μήνα μόνο για το Σέγγεν μιλάω. Και έχω τονίσει πάρα πολύ πόσο σημαντικό είναι το Σέγγεν, ότι είναι δώρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να το ενισχύσουμε ή να το αποδυναμώσουμε. Ε, πολύ σοβαρά μας προβληματίζουν όλες αυτές ε, οι δηλώσεις ε, ε, και είμαστε σε επαφή με το Παρίσι, με τη Ρώμη και με την Κοπεχάγη για να δούμε τι κάνουν και κατά πόσο ανταποκρίνονται όλα αυτά ή δεν ανταποκρίνονται προς το Σέγγεν και τους κανόνες του. Επίσης κοιτούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την αξιολόγηση του Σέγγεν και την εκτίμηση έτσι ώστε εκ των προτέρων να δούμε ε, πώς θα αλλάξει το σύστημα αυτό του ελέγχου μεταξύ ίσων ομοτήμων, αυτό το peer review, ε, μήπως χρειαστεί αλλαγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με αυξημένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χρειαζόμαστε περισσότερα εργαλεία στη διάθεσή μας για να βοηθούμε τα κράτη-μέλη, να ε, είμαστε καλύτεροι στην έκδοση των ε, κατευθυντήριων γραμμών και να δούμε ποιες είναι οι έκτακτες περιστάσεις ε, που μπορεί να οδηγήσουν σε αναστολή για να μην έχουμε μονομερείς δράσεις που διακυβεύουν όλο το σύστημα. Να είστε βέβαιοι ότι θα τονίσω ότι χρειάζεται περισσότερη ευρωπαϊκή συμμετοχή και όχι λιγότερη. Το Δουμπλίνο. Δύο. Βεβαίω συνδέεται με αυτό, αλλά είναι μια παράλληλη διαδικασία και είναι τμήμα των διαπραγματεύσεων του πακέτου για το άσυλο ε, που γίνεται η διαβούλευση αυτή στο Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να διατηρηθεί η ευθύνη του πρώτου του κράτους ε, υποβολή της αίτησης ασύλου, αλλά να μπει και ένας μηχανισμός κατεπήγοντος, έτσι ώστε σε έκτακτες ιδιαίτερες περιστάσεις να μπορεί να αναστέλλεται ο μηχανισμός. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ επίμαχο στα κράτη-μέλη, είναι πάρα πολύ μικρή υποστήριξη για αυτόν τον κατεπήγοντα μηχανισμό και είναι από τα πιο δύσκολα και πιο ακαθόδη σημεία της όλης διαπραγμάτευσης για το πακέτο του ασύλου η λύση του ελληνικού προβλήματος δεν είναι αυτή. Η λύση για την Ελλάδα είναι παράλληλα να στήσει ε, και ένα σύστημα ασύλου και να ισχύει για όλη την Ευρώπη. Αν υπάρχει παντού στην Ευρώπη ένα τέτοιο ε, σύστημα θα μοιράζεται και ε, το άχθος. Να συνεχίσουν οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα δράση στην Ελλάδα και την υποστηρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναλαμβάνω, υποστηρίζουν και τα κράτη-μέλη με πολλά χρήματα, ε, με διερμηνεί, υπαλλήλου, πραγματοκρομοσύνη, για να βοηθήσουν την Ελλάδα να στήσει ένα σύστημα ασύλου που να ευθυγραμμίζεται με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Έχουν γίνει πολλά, αλλά απομένουν ακόμα πολλά να γίνουν. Αλλά όλα αυτά γίνονται παράλληλα με τι διαπραγματεύσει για το σύστημα του ασύλου. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για όλες τις απαντήσεις που δώσατε. Περνάμε στις υπόλοιπες ερωτήσεις προς τον Επίτροπο Άντορ. Κανονικά έχουμε 20 λεπτά για κάθε επίτροπο. Δυστυχώ δεν θα προλάβουμε να καλύψουμε όλες τις ερωτήσει. Η πρώτη ερώτηση προς τον Επίτροπο Άντορ είναι υπαριθμό 13 του κυρίου Φρεντερικ Νταρντέν για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Η κυρία Μπέρες αντεκαθιστά εδώ τον κύριο Νταρντέν. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, σας είμαι ευγνώμων για το ζωηρό ενδιαφέρον που δείξατε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Φέτος ε, θα είναι κρίσιμη χρονιά για το μέλλον του Ταμείου, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να καταθέσει πρόταση για τους ε, κανόνες και τις διατάξεις που διαπούν το Ταμείο και τον τρόπο λειτουργία του στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Του τελευταίου μήνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβησε διαβουλεύσεις για τα, για το, στους πιο σημαντικούς ενδιαφερόμενους και μετόχους του Ταμείου. Ε, παρακολουθήσαμε και εξετάσαμε διεξοδικά την ε, ε, έκθεση πόρτας για το ταμείο αυτό που ε, εξέτασε το Κοινοβούλιο πριν από μήνες και μετά από την εμπειρία που συλλέξαμε από την παρούσα μορφή του Ταμείου και από τα πορίσματα των διαβουλεύσεων έχουμε βάσιμες ελπίδες ότι η τελευταία πρόταση θα βελτιώσει αισθητά το Ταμείο και τη λειτουργία του μετά το 2013 και θα επιλύσει κυρίως δύο προβλήματα από τον υπάρχοντα μηχανισμό χρηματοδότησης. Το πρώτο θέμα είναι ο χρόνος που χρειάζεται από τη στιγμή χορήγηση μια βοήθεια ε, από τη στιγμή που έχει υποβάλει σχετική αίτηση ε, ένα κράτο. Γιατί είναι χρονοβόρη διαδικασία εξέταση μια τέτοια έταση. Θέλουμε να βρούμε τρόπου για να διευκρινίσουμε να πλουστεύσουμε τι πληροφορίε που θα οφείλει να καταθέσει ένα κράτο για να αποδείξει ότι είναι επιλέξιμο το αίτημά του για χρηματοδότηση. Πολύ ε, χρονοβόρα είναι και η διαδικασία για την απόκτηση της έγκρισης μιας αίτησης από τα δύο σκέλη της Δημοσιονομικής Αρχής. Έτσι καθυστερούν οι πληρωμές και αυτό που βαίνει βάρος ε, των ε, δικαιούχων γιατί δεν ε, είναι πρόθυμα τα κρατη να δώσουν κονδύλια για τις προσλήψεις, για την απασχόληση κτλ. Οπότε έχουν αυξηθεί αισθητά οι αιτήσει για χρηματοδότηση από το Ταμείο τα τελευταία δύο χρόνια και αυτό ε, καθιστά πιο δύσκολο τον εντοπισμό συγκεκριμένων περιθωρίων από τα οποία θα αντιλήσουμε τις ε, εισφορέ. Η έγκριση της χρηματοδότησης για το 2011 έπρεπε να αναβληθεί για πρώτη φορά γιατί δεν είχαμε αρκετές πιστώσεις πληρωμών και άμεση διάθεσή του. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε κι εσείς ότι δεν βοηθάει τους ε, εργαζόμενους που έχασαν τη δουλειά τους και χρειάζονται άμεσα μία βοήθεια. Θα πρέπει να βρούμε λύσει στα προβλήματα αυτά και να βρούμε το, ένα μηχανισμό χρηματοδότησης του Ταμείου που θα συνάδει με τους, με τους στόχους που έχουμε. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις αυτή τη στιγμή που εξετάζονται. Για παράδειγμα, το Ταμείο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ή όχι, ή θα μπορούσε να έχει δικό του προπολογισμό ή και όχι. Μέχρι στιγμή δεν έχει ληφθεί απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο για να αντιμετωπιστούν τα θέματα, αλλά το φθινόπωρο θα καταθέσει προτάσει για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή ε, στην Παγκοσμιοποίηση, λαμβάνοντα υπόψη το συμφέρον των ε, εργατών και εργαζομένων πρώτα απ' όλα. Και περιμένω τώρα και τι δικέ σα απόψει. Σα ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τρει ε, συμπληρωματικέ. Πρώτα κυρία Μπερέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εκ μέρους του κυρίου Ντερντέν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την απάντηση που δώσατε. Εμείς ε, φυσικά θα υποστηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία που θα επιταχύνει τη διαδικασία για να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους ε, που απολύθηκαν είτε εξαιτία της παγκοσμιοποίησης είτε εξαιτία της κρίσης. Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε δύο δυσκολίες. Η πρώτη δυσκολία έγκυται στο χαρακτήρα στήριξης προς εργαζόμενους που θα πρέπει να παραμείνει ε, ύψιστη προτεραιότητα. Με την αναθεώρηση των διαδικασιών δεν θα πρέπει το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση να μετατραπεί σε ένα ακόμη μηχανισμό ε, μιας πολιτικής συνοχής. Γιατί τότε όλα τα κοινοτικά κονδύλια πέραν της εξωτερικής πολιτικής ή της ε, έρευνας και ανάπτυξης θα χαρακτηρίζονται ως πολιτική συνοχής έχουμε ιδιαίτερου στόχου και θα πρέπει να έχουμε και ιδιαίτερου μηχανισμού. Και ένα τέτοιο μηχανισμό ξεχωριστό θα πρέπει να είναι το, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Θα ήθελα να συνεννοηθείτε με του ε, επιτρόπου με τους άλλους επιτρόπους ε, που έχουν αρμοδιότητα σε θέματα ανταγωνισμού ή σε θέματα βιομηχανικής πολιτικής. Ο κύριος Χούντη, συμπληρωματική, μισό λεπτό. Στι αρχές του χρόνου σε σχετική ερώτηση αν η ελλάδα έχει καταθέσει αίτηση για να ενεργοποιηθεί το ευρωπαϊκό ταμείο για την παγκοσμιοποίηση είχατε απαντήσει όχι. αυτή η απάντηση έκανε αίσθηση στην ελληνική πραγματικότητα λόγω της οικονομικής και ε, κοινωνικής κατάστασης που βρίσκεται η χώρα. η ερώτηση που σας κάνω είναι απλή. μετά έξι μήνες έχει καταθέσει η χώρα μου αίτηση για ενεργοποίηση του ταμείου παγκοσμιοποίησης για στήριξη των εργαζομένων που πλήττονται από τη χρηματοοικονομική κρίση; αν ναι αν έχετε αυτή την πληροφορία σας παρακαλώ πείτε μου αν έχει εγκριθεί. αν όχι μπορείτε να εξηγήσετε γιατί δεν κατατίθεται από την ελλάδα τέτοια αίτηση. ευχαριστώ πολύ. Και τέλος η κυρία Χάρκιν. Είχα μία ερώτηση πιο κάτω που δεν θα προλάβουμε να την απαντήσουμε για τα περιθώρια του Γεωργικού Ταμείου και του Ταμείου παγκοσμιοποίηση. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δώσετε ήδη μία απάντηση. Και αν θα συγχωνευτούν τα δύο ταμεία, πιστεύετε θα, θα αυξηθεί ο προπολογισμό του Κοινωνικού Ταμείου εφόσον συγχωνευτεί με το Ταμείο τη παγκοσμιοποίηση. Μιλήσατε για τι δυσκολίε ε, που αντιμετωπίζει η Επιτροπή με τα δύο σκέλη τη Δημοσιονομική Αρχή. Από τη στιγμή που τα κράτη-μέλη υποβάλλουν αίτηση για το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση, δεν θα πρέπει να ξεκινήσουν από μόνα του να θεσπίζουν κάποια μέτρα για τα οποία ζήτησαν τη στήριξη του Ταμείου Παγκοσμιοποίηση, ώστε να μην περιμένουν οι εργαζόμενοι εργάτε εργάτες την εφαρμογή, την κινητοποίηση των κονδύλιων του Ταμείου. Χωρί μικρόφωνο, επίτροπο. Χαίρομαι, γιατί από τη συζήτηση επιβεβαιώθηκαν ε, οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση να συμπεριληφθεί στι επόμενε δημοσιονομικέ προοπτικέ και να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό και ισχυρότερο μηχανισμό για την ε, αρρωγή των εργαζομένων που χάνουν την δουλειά του. Και μάλιστα στην επόμενη περίοδο η δημοσιονομική εξυγίαση θα παραμείνει στο, ως προτεραιότητα του προγράμματος των περισσότερων χωρών μελών και θα είναι πολύ χρήσιμο για τα κράτη-μέλη να υπάρχει ε, ένας ισχυρός μηχανισμός αποτελεσματικός και κοινοτικό που θα βοηθήσει τους εργαζόμενους που χάνουν ξαφνικά τη δουλειά τους. Όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχουν πολλά εκρεμή θέματα σχέση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με το Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Το Κοινωνικό Ταμείο εμπίπτει στην ε, κοινή διαχείριση, ενώ ένα τέτοιο σύστημα δεν συνάδει με τους στόχους του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης. Δεν ξέρω τι μορφή θα βρούμε τελικά, αλλά το θέμα της διαχείρισης θα είναι πολύ σημαντικό, θα είναι κέριο προκειμένου να επηρεάσουμε τις τελικές ρυθμίσεις για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη για ένα ξεχωριστό ταμείο και ανάγκη να ληφθεί υπόψη και το θέμα της ταχύτητας διεκπαιρέωσης ε, μιας αίτησης. Και τώρα, αλλά και κατά πάσα πιθανότητα στο μέλλον, πολλές χώρες μέλη θα προσπαθήσουν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα που θα είναι επιλέξιμα και από το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αυτό που είναι σημαντικό όμως είναι να είναι δυνατή η πρόσβαση όλων των χωρών μελών στο Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, εφόσον προκύψει ανάγκη αντιμετώπιση μια ξαφνική κρίση στην απασχόληση. Η δεύτερη ερώτηση επισήμανε τη δυσκολία του ορισμού της επιλεξιμότητας στον τρέχοντα κανονισμό και αυτό το θέμα το εξετάζουμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα μεγαλύτερο επίπεδο ευκρίνειας, σαφήνειας, αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να επεκτείνουμε τον προσωρινό κανονισμό, να τον επιμηκύνουμε μέχρι το τέλος της περίοδου των δημοσιονομικών προοπτικών σε ό,τι αφορά τους κανόνες για την αντιμετώπιση κρίσης προκειμένου να γίνει το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση πιο αποτελεσματικό αναχαιτίζοντας τις συνέπειες της κρίσης για τους εργαζόμενους. Ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη ερώτηση του κυρίου Χουντή σχετικά με το καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων. Ο Μήπως μπορείτε να μας πείτε πόσες ερωτήσεις θα πάρετε ακόμα μέχρι να ε, ολοκληρωθούν οι εργασίες. Είπα ότι έχουμε 20 λεπτά για κάθε επίτροπο που σημαίνει ότι θα πάμε μέχρι και την ερώτηση την επόμενη την 15 της κυρίας Μπλινκεβιτσούτε. Ίσως, ε, μάλλον δεν θα πάμε στη δική σας, γι' αυτό ίσως μπορείτε να κάνετε μια συμπληρωματική σε άλλη ερώτηση. Για 14, ο Επίτροπος. Ε, πρόεδρε, αγαπητά μέλη, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η ελληνική κρίση έχει υψηλό κοινωνικό κόστος ε, για τους πολίτες στην Ελλάδα. Όμως το κόστος αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα δημοσιονομικών ανισορροπιών, ευθύνουσας ανταγωνιστικότητας, ε, πολλές δυσκολίες που προσπαθούν προσπαθεί να επιλύσει το μνημόνιο. Μερικοί ισχυρίζονται ότι δεν ε, σέβεται το μνημόνιο την αρχή της επικουρικότητας που προβλέπεται στη συνθήκη για τη λειτουργία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό είναι σωστό τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο, όπως σας είπα, καταρτίστηκαν σε στενή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και εγκρίθηκαν από το ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι σεβόμεθα την, αρχική, ε, την αρχή της επικουρικότητας. Ο χάρτης ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζει την άποψή μου. Το άρθρο 28 του χάρτη προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι και οι οργανώσεις τους ε, πρέπει να προστατεύονται και έχουν το δικαίωμα να ε, διαπραγματεύονται, να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις στο κατάλληλο επίπεδο και σε περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων να καταλήγουν σε ε, συλλογικές ενέργειες συμπεριλαμβανομένης και της απεργίας. Όμως το άρθρο 51 του χάρτη λέει ότι οι διατάξεις του χάρτη αφορούν τους οργανισμούς, τους θεσμούς, ε, τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας μόνο εφόσον τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη κοινοτική νομοθεσία που να ρυθμίζει ποια συλλογική σύμβαση υπερισχύει πια όταν οι συμβάσεις συνάπτονται σε διαφορετικό επίπεδο ή όταν πρόκειται για επέκταση των συλλογικών συμβάσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο μέσα από παρέμβαση του κράτους. Άρα δηλαδή αυτά είναι αποκλειστική αρμοδιότητα εθνικών κρατών που σαφώς και σεβόμεθα ε, τις ε, διεθνείς συμβάσεις περί εργασίας. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, θεωρώ ότι απάντησα ικανοποιητικά στην ερώτηση του κυρίου Ευρωβουλευτού. Ε, θεωρώ επίσης ότι σας έπεισα ότι τα δημοσιονομικά και άλλα μέτρα που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο είναι καθοριστική σημασία, είναι κέρια αν η Ελλάδα επιθυμεί να βγει από την κρίση. Και είμαι σίγουρος ότι αρκετοί από εσά ε, θα έχουν ακούσει ότι δεν ισχύει αυτό που λέγεται περί αποτυχίας ε, εφαρμογής επικουρικότητας. Κύριε Χουντή, συμπληρωματική ερώτηση. 30 δευτερόλεπτα. Κύριε Επίτροπε, λυπάμαι ότι για άλλη μια φορά η απάντησή σας δεν ήταν σαφής, γιατί την ίδια περίπου απάντηση μου δίνεται και σε γραπτές ερωτήσεις. Αν πράγματι η Κομισιόν σέβεται ότι το καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων είναι θέμα εθνικής νομοθεσίας, τότε παραβιάζετε ή όχι το ρόλο σας με βάση τις συνθήκες όταν ζητάτε να καταργηθεί ουσιαστικά το καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων. η ερμηνεία που δίνετε δεν την υιοθετούν και τα ευρωπαϊκά συνδικάτα που σας έχουν καταγγείλει για παραβίαση των συνθήκων και η ερώτησή μου είναι ποιος το ζητάει να καταργηθούν οι συλλογικές συμβάσεις εσείς το διεθνές νομισματικό ταμείο οι δανειστές της ελλάδας της πορτογαλίας της ιρλανδίας; σας παρακαλώ ποιο σαφή απάντηση. Ο Επίτροπος. Μικρόφωνο παρακαλώ. πολλές θεσμικές ρυθμίσεις όπως ε, και οι μισθολογικές ε, σε διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχουν τέτοιου τους ρυθμίσεις, αλλά εδώ έχουμε έκτακτες ρυθμίσεις έκτακτης κατάστασης που αντιμετωπίζονται μέσα από πολιτικές που ε, καταρτίζονται από κοινού Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Τομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και κυβερνήσεις ε, των κρατών μιλών. Για αυτά μιλάμε. Πράγματι, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα ανοιχτά ερωτήματα, ορισμένα ετέθησαν και από την Συμφωνία Europlus ε, το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε αρκετές συζητήσεις ε, σχετικά με τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον κοινωνικό διάλογο και την οικονομική, κοινωνικό διάλογο και την οικονομική διακυβέρνηση. Κοινωνικό λοιπόν διάλογο και οικονομική διακυβέρνηση. Συνεχίζεται η συζήτηση. Δεν λέω ότι έχουν απαντηθεί όλα τα εκκρεμή ερωτήματα. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο ανέλαβα την πρωτοβουλία να οργανώσω μία ακρόαση για το πώς ε, ρυθμίζονται θέματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην ακρόαση αυτή θα συμμετάσχουν και οι κοινωνικοί εταίροι και άλλοι εμπλεκόμενοι το Σεπτέμβρη θα λάβει η χώρα αυτή η μερίδα. Θα συνεχιστεί λοιπόν η συζήτηση και ελπίζω εν ευθέτω χρόνο να βρούμε τις κατάλληλες απαντήσεις. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση ε, προς τον κύριο Όντο, αριθμό 15 της κυρίας Βλίνκεβιτσούτε. Ίσως να απαντούσατε σύντομα ε, και εσείς και οι συμπροματικές σύντομες και οι δευτερολογίες σας. 15. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων είναι η θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεμελιώδης μαζί με την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, ε, κεφαλαίων και υπηρεσιών είναι πυλώνας Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει συνεισφέρει τα τελευταία 50 χρόνια στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Βεβαίως έχει και μεγάλη κοινωνική διάσταση γιατί σφυριλατεί την κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ένταξη των μεταναστών, των εργαζομένων ε, και των μελών της οικογένειας τους ε, στη χώρα που τους υποδέχεται. Έχουν το δικαίωμα οι πολίτες της Ένωσης να να κινούνται συγγνώμη, ελεύθερα και προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και των μελών ε, της οικογένειά του. Την 1η Μαγιά του 2011 ήταν σημαντική ημερομηνία για την Ένωση γιατί ε, καταργούνται οι περιορισμοί ε, του δικαιώματος εργασίας των 8 κρατών που μπήκαν το 2004 την Πρωτομαγιά και μπορούν πλέον να εργάζονται ελεύθερα σε όλα τα κράτη-μέλη. Ακόμα εφαρμόζονται προσωρινά μέτρα για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά όταν λήξει η δεύτερη φάση 31 Δεκάτου 2011 ελπίζω να λήξουν και αυτά. Το τέλος των μεταβατικών αυτορυθμίσεων σημαίνει ότι μπορούν περισσότεροι πολίτες της Ένωσης να εκμεταλλευτούν ε, πλήρως ε, την ελευθερία αυτή και να εργαστούν σε άλλη χώρα. Αυτό διανοίγει μεγάλες ελευθερίες και ευκαιρίες για τα ε, πρόσωπα και για την οικονομία. Γνωρίζω ότι η κινητικότητα και η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων είναι σημαντικά και για το κοινοβούλιο σας. Το Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για την προώθηση της κυκλοφορίας των εργαζομένων και με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον περιμένει την περαιτέρω συζήτηση. Γνωρίζουμε όμως ε, ότι παρά τη μεγάλη κοινοτική νομοθεσία στον τομέα αυτό, πολλοί πολίτες θεωρούν ότι παραμένουν πολλά τα εμπόδια για να εργαστεί κανείς σε άλλο κράτος μέλος. Επανειλημμένα και πρόσφατα έχει εκφραστεί αυτό. Η έκθεση Μόντι της 9 η Μαΐου του 2010, μια νέα στρατηγική για την εσωτερική αγορά, τονίζει ότι είναι γενικά επιτυχής η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από πλευράς νομικής, αλλά δεν χρησιμοποιείται, είναι η λιγότερο χρησιμοποιούμενη από τις τέσσερις ελευθερίες. Χρειάζεται ε, πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή Η επιβολή αυτής της ελευθερίας ε, είναι σημαντική και φαίνεται ότι υφίστανται διακρίσεις ακόμα οι πολίτες της Ένωσης με βάση την εθνικότητά τους και θα πρέπει να προστατεύονται με σωστό τρόπο. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αξιολογούν τώρα και εξετάζουν την κοινοτική νομοθεσία για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, ιδιαίτερα τον κανονισμό 16-12 ε, του 68 και ε, ελέγχουν και εξετάζουν κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί ε, η ελευθερία αυτή και αν χρειαστεί να καταθέσουμε και πρωτοβουλία το 2012. Έρχεται λοιπόν η πρωτοβουλία αυτή πολύ επίκαιρα και θα το συζητήσουμε για να δούμε ποια περαιτέρω δράση πρέπει να επιλεγεί για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, η κυρία Μπλίνκα Τσούτε. Αν κάνετε σύντομη ερώτηση και απαντήσει ο κύριος Άντορ, Γιατί ε, έχουμε περάσει στο χρόνο του Επιτρόπου κυρίου Χάν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κανονισμός που μας είπατε θα βελτιωθεί και θα αναθεωρηθεί ε, το 2012. Θα ήθελα όμως να μου πείτε το εξής, το εξής ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο τα θετικά αξιολογεί, τα αρνητικά δεν τα αξιολογεί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Παράδειγμα, Πολλοί εργαζόμενοι έφυγαν από τη χώρα τους, άνθρωποι με προσόντα, ειδικευμένοι, ε, πολύ αξιόλογοι και πήγαν να εργαστούν σε άλλα κράτη-μέλη. Δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ταμείο αποζημίωσης των κρατών που εκπαίδευσαν αυτούς τους εργαζομένους και στη συνέχεια χάνουν αυτό το εργατικό δυναμικό που είναι αξιόλογο και ειδικευμένο. Κύριε Πρόεδρε, απαντά Επίτροπος. Όντως είναι εύστοχο το ερώτημα και πρόσφατα έγιναν πολλές συζητήσεις για τη Βρωτομαγιά. Το συζήτησα με υπουργού εργαζο... ε, απασχόλησης των χωρών Βίσεγκράτ, των χωρών της Βαλτικής και βεβαίως εξετάζουμε και διερευνούμε κατά πόσο ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις. Ιδιαίτερα αφορά ορισμένα επαγγέλματα όπου η ελεύθερη κυκλοφορία δεν οδηγεί σε ένα κυκλικό φαινόμενο αλλά σε διαρροή εγκεφάλων σε ένα μονόδρομο. Όταν παρατηρούνται τέτοιες ε, τάσεις εναπόκειται κυρίως στις κυβερνήσεις των χωρών αυτών ε, για ε, αντίστοιχες ευκαιρίες, εκπαίδευση, αμοιβή ε, ευκαιρίες για απασχόληση. Αφορά ιδίω τα ιατρικά επαγγέλματα αυτό και θα πρέπει να διευκολύνεται ακριβώς η παραμονή ε, των εργαζομένων στη χώρα τους. Ε, θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε, να παρακολουθούμε αυτό το πρόβλημα και θα το συζητήσουμε με τις εν λόγω κυβερνήσεις όπως και στο παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ. Οι επόμενε ερωτήσει θα απαντηθούν γραπτό. Σα ευχαριστώ όλους και τον κύριο Όντορ. Και ερχόμαστε σε ερωτήσει προς τον κύριο Χάν. Πρώτη ερώτηση για τον κύριο Χάν Πέτερ Μάρτιν. Ανακατανομή των χρηματοδοτικών μέσων του Περιφερειακού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής. Όποτε είναι έτοιμος. Επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ευθύ εξ αρχή ότι από το τίτλο ε, των Διαρθωτικών Ταμείων για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο από το 2007 ως το 2013 στα πλαίσια ε, των προγραμμάτων των επιχειρησιακών που είναι πάνω από 400 έχουν ήδη κατανεμηθεί οι πόροι. Μαζί με τις περιφέρειες και τα κράτη-μέλη έχουν συμφωνηθεί αυτό είναι τμήμα της συνολικής διαδικασίας στην αρχή μιας προγραμματικής περίοδου. Το συζητούμε με τις κυβερνήσεις, με τα κράτη-μέλη και με τις περιφέρειες και συμφωνούμε τα προγράμματα για όλη την προγραμματική περίοδο για να ορίσουμε και τη χρηματοδότησή τους και την πρικοδότησή τους για όλη την περίοδο για την κοινή διαχείριση και τη διοίκηση αυτών των προγραμμάτων και αρμόδια είναι τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες ή οι περιφέρειες μαζί με τα κράτη για την επιτόπου εφαρμογή και για την επιλογή των προγραμμάτων και για την εκτέλεσή τους και για τον έλεγχο τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο. Είναι αρμόδια ε, τα κράτη ή οι περιφέρειες. Ήδη από την αρχή της παρούς περίοδου το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας και της πρόθεσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ήταν σημαντικό και παραμένει προτεραιότητα στην περιφερειακή πολιτική εξού και... Ε, έχουμε μέτρα και συγκεκριμένες προσφορές σε πολλά από τα 400 αυτά προγράμματα. Γενικά στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, μετά από τη συμφωνία με τις περιφέρειες και τα κράτη-μέλη, ο προϋπολογισμός είναι 9,2 δισεκατομμύρια ευρώ για μια υφόρο ενεργειακή πολιτική με κέντρο βάρους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βελτίωση της εξοικονόμησης και της απόδοσης της ενέργειας. Και μετά από απόφαση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου του 2009 δημιουργήσαμε επιπλέον τη δυνατότητα μέχρι 4% των πόρων του Ταμείου για την Ανάπτυξη, την Περιφερειακή, να πηγαίνουν εκεί για τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης ενέργειας ε, σε ε, θέματα κτηρίων και κατοικιών. Και περίπου τα μισά κράτη-μέλη έχουν κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας ήδη. Αλλά πρέπει να σας πω ότι η Γαλλία ε, πραγματικά ε, έχει προχωρήσει σε αυτή τη ε, ε, χρήση, αυτή τη δυνατότητα. Ευχαριστώ. Κύριος Μάρτιν. Ευχαριστώ. Κύριε Πίτροπε, μην με παρεξηγείτε, αλλά για να είμαι σοβαρή. Ε, ε, σας κάνω την ερώτησή μου. Είναι Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 10% των 51 δις που χρησιμοποιούν σήμερα για χρηματοδότηση νέων ε, δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Πολλά μας είπατε και πολύ σωστά, αλλά δεν σας ρώτησα εγώ αυτό. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα και να πούμε ότι μάλιστα καταλάβαμε. Μάλιστα βγάζουμε τα συμπεράσματα από τη Φουκουσίμα και παίρνουμε σοβαρά υπόψη το 2020 και για να γίνει αλλαγή και στην ηλεκτρική ενέργεια θα πρέπει το ρεύμα από τη Βόρεια Γερμανία να φτάσει στην Αυστρία. Ε, ε, ακούσατε ε, τι γίνεται. Έχετε και εμπειρία από τα ηλεκτρικά εργοστάσια. Για να φτάσει κάπου το ρεύμα χρειάζονται δίκτυα, καλώδια. Θα χρηματοδοτήσετε αυτά. Γιατί είναι επίγον να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια και όχι αυτά που αποφάσισαν οι προ-προκάτοχοί σας, ο Επίτροπος. Ναι, διάβασα πολύ προσεκτικά την ερώτησή σας και σας έδωσα μια πολύ ακριβή απάντηση με βάση τους κανόνες που ισχύουν για την περιφερειακή πολιτική. Και η ουσία της πολιτικής αυτής είναι ότι μαζί με τα κράτη-μέλη συμφωνούμε την πολιτική αυτή. Αυτές οι συμφωνίες δεν μπορούν να καταγγελθούν μονομερώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε από τις περιφέρειες, ούτε να αλλάξουν. Και εγώ προσωπικά θα χαιρόμουν και θα επιθυμούσα ήδη από τώρα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας να χρησιμοποιούνται. Εγώ τρέχω από διάσκεψη σε διάσκεψη, από χώρα σε χώρα, ε, ως ε, ζωντανός ε, ε, ζωντανή απόδειξη όλων αυτών η αύξηση ε, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι από τα κέντρα βάρους για την πολιτική του 2020. Θεωρώ ότι θα υπάρξει υψηλότερη χρηματοδότηση και στην ε, περιφερειακή πολιτική για τον τομέα αυτό και σίγουρα ε, με τον συνάδελφο Oettinger θα ε, συζητήσουμε και για επενδύσεις στα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών και για τα δίκτυα ε, παροχής ενέργειας. Εάν σήμερα οι περιφέρειες ε, έχουν τη δυνατότητα ε, μεταφοράς πιστώσεων από τις υπάρχουσες πιστώσεις, σίγουρα είμαστε πολύ πρόθυμοι να το συζητήσουμε και να τους δώσουμε τη δυνατότητα αυτή να κάνουμε σοβαρές συζητήσεις. Αλλά επαναλαμβάνω, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούμε μόνο μερός να αλλάξουμε αυτές τις συμφωνίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η επόμενη ερώτηση είναι η παριθμόν 20 της κυρίας Είναι εκπλήρωση των στόχων στον τομέα των πληρωμών των διαρθρωτικών ταμείων. Ο Επίτροπος Χάν. Κυρία ε, Βουλευτή, ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Όσον αφορά το θέμα του ποσοστού απορρόφησης ε, και την αναγνώριση αυτού για την εκταμείευση κοντιλίων, ε, θα ήθελα ήδη τώρα να σας παραπέμψω στους ισχύοντες κανονισμούς ε, σχετικά με το ανώτατο όριο της χορήγης κοντιλίων. Λέξη κλειδί εδώ είναι το περίφημο capping. Υπάρχει δηλαδή ένας κανόνας που λέει ότι για να υπάρξει μια συγκεκριμένη κλίμακα ανακράτος μέλος λαμβάνεται υπόψη ένα συγκεκριμένο ποσό που είναι σε αναλογία και σε συνάρτηση με το ΑΕΠ της χώρας και η ετήσια χρηματοδότηση δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει αυτό το ανώτατο όριο. Ε, κατά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα σκεφτούμε κατά πόσον αυτό το ανώτατο όριο είναι αιτιολογημένο ή όχι, μήπως χρειάζονται προσαρμογές, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη δυνατότητα απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Όσον αφορά την επίτευξη των στόχων, να σας ε, παραπέμψω στο ε, στην πέμπτη έκθεση περί συνοχής ε, και στη αναθεώρηση του προεπολισμού που αναφέρεται ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν και πάρα πολλά προγράμματα, το σύστημα των κινήτρων, το σύστημα των στόχων αναφέρονται όλα αυτά τα οποία έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα καταθέσει για την πολιτική μετά το 2014. Όσον αφορά το ε, ποσοστό σφάλματος, ε, νομίζω έχω τοποθετηθεί επανειλημμένα και εδώ ε, σας έχω μιλήσει για την αναθεώρηση των πολιτών προγραμμάτων και σας έχω πει ότι πράγματι ε, υπάρχουν κονδύλια τα οποία δαπανώνται για πολιτή προγράμματα και το ελεγκτικό συνέδριο ελέγχει την εφαρμογή ενός προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια ενός και μόνο έτους. Άρα δηλαδή καθαρά μεθοδολογικά προκύπτουν προβλήματα, προκλήσεις πέστετες, γιατί στο πλαίσιο της ε, περιφερειακής πολιτικής υπάρχουν τρία επίπεδα ελέγχων. Υπάρχει ο ετήσιος έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά ε, αυτός ξεκινάει μετά το πρώτο επίπεδο ελέγχου. Άρα δηλαδή θα υπάρχει πάντα στην αρχή μεγαλύτερο ποσοστό σφάλματος από ότι στο τέλος του κύκλου ζωής του προγράμματος. Παρόλα αυτά ε, η προκάτοχός μου, η κυρία Χούπνερ, ε, κατάρτισε μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα πρόγραμμα δράσης ε, το οποίο πράγματι αποδείχθηκε αποτελεσματικό. Και ένα από τα μέτρα που προτάθηκαν ήταν η, γενική, η αρμόδια γενική διεύθυνση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να αναστείλει τις πληρωμές κατά το μέγιστο μέχρι και έξι μήνες. Αυτό το εργαλείο ε, χρησιμοποιήθηκε την προηγούμενη χρονιά για πάνω από 50 φορές και οι αναστολές ε, πληρωμών πριν περάσουν οι έξι μήνες ε, ήρθησαν και επανελήφθησαν οι χρηματοδοτήσεις γιατί δεν υπήρχαν πλέον προβλήματα. Σας παρακαλώ όμως όπως σας είπα στο ποσοστό σφάλματος να λαμβάνετε υπόψη σας ότι η περιφερειακή πολιτική είναι διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ορισμένα πράγματα να είναι καθαρά θεωρητικά και στην πρακτική τους εφαρμογή να ελέγχονται ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Ε, το θέμα ε, των ε, κρατικών και δημόσιων συμβάσεων. Αυτό το συζητάμε με πολλά κρατημέλη, με τους τελικούς αποδέκτες οι ε, δημόσιες συμβάσεις και οι δημόσιοι διαγωνισμοί λαμβάνουν και κατέχουν το 70% του ποσοστού σφάλματος. Κατόπιν τούτου με τον κύριο Μπαρνιέ είπαμε ότι πρέπει να απλουστεύσουμε λιγάκι το σύστημα για να υπάρξει και χαμηλότερο ποσοστό σφάλματος. Αν θέλετε δηλαδή σε αυτό τον τομέα προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, να εξελιχθούμε περαιτέρω. Ευχαριστώ κυρία Γένσεν. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την ε, πληρέστατη και εξαιρετική απάντηση που δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα αυτά τα προβλήματα που δυστυχώ δεν έχουν μειωθεί με την οικονομική κρίση γιατί έχουν αυξανόμενε δυσκολίε εξασφάλιση χρηματοδότηση τα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω τι θα σημαίνει αυτό για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Η στήριξη των διορθωτικών ταμείων οδηγεί τελικά σε ανάπτυξη των περιφερειών. Είναι ορατά τα αποτελέσματα και έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άλλες προτάσεις, άλλες ιδέες ε, για το πώς θα κάνει πιο αυστηρό την παρακολούθηση και την εκπλήρωση των στόχων και των αναπτυσσιακών για να διαπιστώνουμε αν πραγματικά τα διάφορα προγράμματα έχουν και αυτά αποτελέσματα. Ο δεδηλωμένος στόχος μας είναι κατά την επόμενη περίοδο, όταν θα εφαρμοστούν τα προγράμματα, τη διαρθρωτική πολιτική να την προσαρμόσουμε στο βαθμό του δυνατού στην στρατηγική μας Ευρώπη 2020. Άρα δηλαδή υπάρχουν ε, βασικοί στόχοι, υπάρχουν προτεραιότητες και όλα αυτά θα προσαρμοστούν στις διάφορες περιοχές όπου βέβαια το καθήκον των περιοχών είναι αν θέλετε, από έναν ε, κατάλογο εστιατορίου, ας το πούμε έτσι, να επιλέξουν κάποια προγράμματα και μετά όμως αφού επιλέξουν τα προγράμματα αυτά, να συζητήσουν μαζί μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να θέσουν ρεαλιστικούς, ποσοτικά μετρήσιμους στόχους, έτσι ώστε από κοινού να καταλήξουμε ε, σε μια συμφωνία συνεργασίας. Αν γίνουν όλα αυτά, στο τέλος της περίοδου θα μπορούμε να δούμε πάρα πολύ καλά κατά πόσον οι στόχοι που από κοινού θέσαμε έγιναν, ε, επιτεύχθηκαν ή όχι. Και αν δεν έχουν επιτευχθεί, να έχουμε τη δυνατότητα και πάλι από κοινού να αναζητήσουμε τα αίτια της αποτυχίας. Ε, οι παράγοντες, τα αίτια που οδήγησαν στην αποτυχία ήταν εσωτερικά ή εξωτερικά. Και αφού γίνουν όλα αυτά, θα εξάγουμε τα συμπεράσματά μας και για, την, ε, για τον περαιτέρω ε, προγραμματισμό. Αυτά λοιπόν ε, είναι μια πολύ σημαντική περαιτέρω εξέλιξη της περιφερειακής πολιτικής κατά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ο κύριος που απουσιάζει. Κύριε Τσικάου, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά η ερώτησή σας απαιτεί διεξοδικότατη απάντηση. Συνήθω τέτοιε ερωτήσεις έχουμε στην... Ε, όχι την ώρα των ερωτήσεων. Καλύτερα να λάβετε γραπτό απάντηση στην ερώτησή σας, οπότε ολοκληρώνεται η ώρα των ερωτήσεων. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο και τους Διερμήνες.